οι διορισμοί αυτοί θα υιοθετηθούν. Η αρμόδια επιτροπή έχει παρουσιάσει μια διόρθωση σε σχέση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτή υιοθετήθηκε σε δεύτερη ανάγνωση και αυτή θα δημοσιευθεί στα πρακτικά καθώς και στο site του ίντερνετ. Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 το διορθωτικό αυτό θεωρείται εγκεκριμένο αν εντός 48 ώρων μια πολιτική ομάδα ή 40 βουλευτές τουλάχιστον ε, το ζητήσουν να ψηφιστεί. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν θα ακολουθήσουμε. Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη και στο επόμενο σημείο αυτής. Έχετε λάβει το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης που έχει εγκριθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της της 17 ε, Σεπτεμβρίου 2009 σύμφωνα με το άρθρο 137 του κανονισμού.